Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Ας αρχίσουμε. Πριν περάσουμε στις ψηφοφορίες, να σας πω στις ανακοινώσεις του Πρόεδρου τι αποφάσεις πήραν χτες οι συντονιστές Πρώτον, ορισμός εισηγητών και συντακτών γνωμοδοτήσεων. Θα σας διαβάσω έναν μεγάλο τίτλο, το μεγαλύτερο που έχει ποτέ σκεφτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για πρόταση, για απόφαση του Συμβουλίου όσον αφορά τη Συμφωνία για τις αεροπορικές μεταφορές και τη Συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών Ισλανδία, ε, Νορβηγία. Οι συντονιστέ σκέφτηκαν επειδή είναι τόσο μεγάλο ο τίτλο, θα πρέπει να είναι ο πρόεδρο που θα αναλάβει αυτή την έκθεση. Αυτή είναι η συνήθι διαδικασία. Αερομεταφορές τώρα. Συμφωνία με την Ελβετία. Ορισμός εισηγητή. Σύμφωνα με το εκπεριτροπής σύστημα που έχουμε με τις πολιτικές ομάδες, το αναλαμβάνουν οι φιλελεύθεροι, Άλντε. Αεροπορική συμφωνία επίσης με τη Βραζιλία τώρα. Οι συντονιστές είπαν ότι αναλαμβάνει η συγγύτρια κυρία Τίκαου. Γνωμοδοτήσεις. Πρόταση για οδηγία που αναδιορθώνει το ευρωπαϊκό πλαίσιο όσον αφορά την φορολογία ενεργειακών προϊόντων για ηλεκτρισμό. Είπαμε θα γίνει γνωμοδότηση. Μετά την αναθεώρηση μάλιστα των αποφάσεων όσο έχουν να κάνουν με τα State Aid Rules, είπαμε ότι τη γνωμοδότηση την αναλαμβάνει η ΓΚΟΕ. Η ΓΚΟΕ δηλαδή βρέθηκε πάνω πάνω στον κατάλογο τώρα Και αυτό συνδυάστηκε με το σημείο 12 που είναι η ανακοίνωση για την ευφύ ενέργεια, smart energy. Η Γκουε κάνει και αυτή την γνωμοδότηση πάντα βάσει του συστήματος εκπεριτροπής. Στη συνέχεια, έκθεση για την λειτουργία και τη ρύθμιση για τα άτομα με αναπηρίες όταν ταξιδεύουν αεροπορικός υπάρχει ανακοίνωση για την εφαρμογή του κανονισμού 261. Οι συντονιστές αποφάσισαν να ζητήσουν άδεια για έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας που να καλύπτει την έκθεση για τα δικαιώματα PRM αλλά και τα δικαιώματα των επιβατών. Η ομάδα σειρά είπε ότι ίσως ήταν καλύτερα να χωρίσουμε τα δύο θέματα, αλλά οι συντονιστές τελικά συμφώνησαν να εξεταστούν μαζί Οπότε θα ζητήσουμε έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας γι' αυτό. Συμφωνήσαμε επίσης να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή ε, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να ετοιμάσουν και εκείνη έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας και ίσως να έχουμε και μία κρόαση από κοινού μαζί τους για τα δικαιώματα των επιβατών. Αυτό θα το δούμε όμως αργότερα βάσει της γνωμοδότησης του εισηγητή και της απόφασης που θα λάβουν οι συντονιστές. Το προσωπικό της Επιτροπής τώρα ετοιμάζει ένα έγγραφο αξιολόγηση της εφαρμογής των μέτρων που έχουν ληφθεί για την εποπτεία των ε, αεροσκαφών. Εδώ δεν έχει αναλυφθεί καμία πρωτοβουλία. Έπειτα έχουμε την ανακοίνωση της Επιτροπής για έναν κοινό χώρο αεροπορικών μεταφορών με τη Μολδαβία. Εδώ αποφασίστηκε να οριστεί εισηγητής και βάσει του συστήματος εκπεριτροπής πάντα η ομάδα ECR αναλαμβάνει αυτήν την ε, γνωμοδότηση. Γνωμοδότηση 11. Ανακοίνωση της Επιτροπής για μια στρατηγική ενεργή χώρου από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ορισμός εισηγητή Βέβαια η Ήτρε αποφασίζει για την ε, αρμόδια επί της ουσίας, αν αποφασίσει για έκθεση πρωτοβουλίας και θα το αποφασίσει αύριο στις 25 του μηνός. Ανάλογα με αυτό λοιπόν θα ε, κάνουμε και εμείς. Αν δεν το κάνουν εκείνοι θα δούμε τι θα κάνουμε εμείς. Ανακοίνωση τώρα για την ε, πράξενη αγορά. Δεν έχουμε εδώ πέρα τίποτα, δεν θα κάνουμε τίποτα. Αυτό αποφάσισαν οι συντονιστές. Το ίδιο και με το έγγραφο εργασίας για τις κλιματικές αλλαγές. Υπάρχει και ανακοίνωση για τους κρατικούς κανόνες. Εδώ πάλι αποφασίσαμε να μην κάνουμε καμία γνωμοδότηση. Επίσης, από την Επιτροπή Αναφορών μου ζητήθηκε κάτι για το air conditioning όταν ε, βρίσκονται σε στάση τα σκάφη. σε αυτούς του... Μας ζητήσαν να πούμε ότι θα έπρεπε να είναι... Η... Όχι στα σκάφη, συγγνώμη, στα φορτηγά, ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό ακόμα και όταν σβηστεί η μηχανή τους. Η απόφαση των συντονιστών είναι για σύσταση να στείλουμε επιστολή στην Επιτροπή Αναφορών λέγοντας ότι όταν λειτουργεί το air conditioning, όταν είναι σταματημένο το φορτηγό, είναι κάτι το οποίο ήδη ισχύει για πολλά καινούρια φορτηγά και θα μπορούσε να γίνει και μια σχετική προσαρμογή σε παλιότερα φορτηγά. Οπότε θα έχουμε προφορική τροπολογία στην έκθεση ΚΟΧ για την οδική ασφάλεια από αυτού. Για την επιτροπολογία τώρα. Ε, αντιρρήσεις όσον αφορά τις ρυθμίσεις και την εποπτεία των αδειών των ε, πιλότων. Ο κύριος Ελκαντράου είναι ο εισηγητής και είπε ότι το μέτρο αυτό δεν έχει πάει ακόμα στο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον τον Ιούλιο. Πριν όμως ε, αντιτεθούμε με την προθεσμία τους τρεις μήνες και τις προθεσμίες μετάφρασης κτλ. Οι συντονιστέ αποφάσισαν να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες από την Επιτροπή και να το ξανασυζητήσουμε το θέμα αργότερα, όταν η ανακοίνωση αυτή μας έχει φτάσει. Στα διάφορα για τα προγράμματα ΣΤΟΑ που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η Γραμματεία ζήτησε να διευκρινίσουμε κάτι για την ε, οικολογική απόδοση και για τις βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιεί η βιομηχανία όσον αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα. Και για μελέτες όσον αφορά το 2011 υπάρχει επιστολή προς το Πρόεδρο για μη πλήρης ε, οι προτάσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα και αποφάσισαν οι συντονιστές για τα εξής. Οι πολιτικές ομάδες πρέπει να υποβάλουν ό,τι οι σχέδια θέλουν για το 2011 για να καλυφθεί ο προπολογισμό του 2011, ώστε να μπορέσουν οι συντονιστέ να αποφασίσουν στι 20 Ιουνίου, στην επόμενη συνεδρίασή μα. Δηλαδή, η προθεσμία για τι προτάσει των πολιτικών ομάδων προ τη Γραμματεία είναι η 6η Ιουνίου του 2011. Κοντεύω, κοντεύω. Ατυχήματα στο Ρήνο. Ήταν απογοητευτική απάντηση του Επιτρόπου στην επιστολή του Προέδρου όσον αφορά τα ατυχήματα στο Ρήνο για το TMS Waldorf και οι συντονιστές αποφάσισαν να ζητήσουν από τον Επιτροπό για την αυσιπλοεία να έρθει εδώ και να μας παρουσιάσει την έκθεση και τα συμπεράσματα όσον αφορά τα ατυχήματα αυτά. Το θέμα τώρα των δύο φίλων και το mainstreaming. Έχουμε πάρει ερώτημα από την Επιτροπή Γυναικών να δούμε πώς έχει το θέμα αυτό μέσα στο Κοινοβούλιο και για τη δουλειά δηλαδή των επιτροπών που γίνεται μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι γίνεται με την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων στις εργασίες αυτές. Η κυρία Τικάου, η αντιπρόεδρό μας που είναι υπεύθυνη για θέματα ισότητας των δύο φύλων, υπέβαλε ένα σχέδιο απάντησης και ζήτησε από τις πολιτικές ομάδες να απαντήσουν αν έχουν σχόλια στη γραμματεία, αν θέλουν κάποια αλλαγή. Η προθεσμία είναι η 1η Ιουνίου γι' αυτό. Συμμετοχή των Πρόεδρων των Επιτροπών σε αντιπροσωπείες ε, πέρα της ποσόστος της αιτήσιας που έχουν διάφορες επιτροπές. Ε, ο κ. Γκρός από το ΕΛΚ το έθεσε και οι συντονιστές αποφάσισαν να ζητήσουν τη συμμετοχή των Πρόεδρων των Επιτροπών ε, εκτός ποσόστοσης βάσει απόφασης που θα παίρνει το Προεδρείο. Τέλος, ο προπολογισμό και το 2012 αποφασίστηκε με βάση των σχεδίων και των προτάσεων για δράσεις και θα προταθεί στις, μέχρι τις 3 Ιουνίου στην Επιτροπή Προπολογισμών. Οι συντονιστές αποφάσισαν βάσει της πρότασης του κ. Λιμπεράτσκη, του εισηγητή και των σχεδόν εισηγητών, αποφάσισαν για τις εξής τρεις προτάσεις πολιτιστική κληρονομιά, ε, μεταφορές και interface όσον αφορά τους διάφορους τρόπους μεταφορών και πρόσβαση για όλους. Αυτά όσον αφορά την συνάντηση των συντονιστών χτες. Κύριε Κράμερ. Στα διάφορα υπάρχει ένα λάθος. Το 2010 στην ΣΤΟΑ είχαμε ζητήσει να εγκριθεί μελέτη και εγκρίθηκε κιόλας για Eco Efficient Transport και στο τέλος δεν λέει για την ένταξη ηλεκτρικών αυτοκινήτων αλλά ηλεκτρικής κινητικότητας που σημαίνει και, άλλων τύπο, και άλλων τύπων οχήματα. Μάλιστα ναι, εντάξει θα το διορθώσουμε λέει ο πρόεδρος το vehicles για την συνάντηση των συντονιστών. Έχει κανείς άλλα σχόλια. Όχι, λοιπόν, εγκρίνονται τα πρακτικά αυτά και θα προχωρήσω στο επόμενο θέμα, δηλαδή τις ψηφοφορίες. Παρακαλώ τοποθετήστε και ελέγξτε ότι είναι τοποθετημένες οι κάρτες σας στην ε, κατάλληλη σχισμή. Κάνουμε τώρα πρώτα μια δοκιμή, αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας. Μήπω έχει κανείς κάνει τίποτε πονηρό. Όχι, όλοι ήσασταν εντάξει. Λοιπόν, προχωρούμε τότε στην πρώτη ψηφοφορία για το σχέδιο συστάσεως για τη δεύτερη ανάγνωση για την κοινή θέση του Συμβουλίου για διαμεθοριακές ανταλλαγές πληροφοριών για θέματα παραβιάσεων και τροχαίων αδικημάτων. Η κυρία Γιάννα Σέντερ, δηλαδή. Τροπολογία 30, Λίχτενμπεργκερ, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29. Εκπίπτει. Το ίδιο 46. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 51 είναι ταυτόσιμου περιεχομένου Βαντάλεν Μπαχ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 του κ. Ρικέ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για την 55 επειδή έχουμε εγκρίνει ήδη την 17 ψηφίζουμε μόνο τις λέξεις τουλάχιστον, at least και μετά το δεύτερο κομμάτι που λέει για τις δυνατότητες απόκτησης νομικής βοήθειας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 του κύριο Ρίκε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 προφορική τροπολογία της κυρίας Σαβισάρ και του κυρίου Μπαχ αντικατάσταση αντί Ο... απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 Λίχτενμπέργκερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και 59. Εκπίπτει. 19. Εισηγητρίας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62 του ε, και του κυρίου Δανέλη να ψηφιστούν μόνο ορισμένε λέξεις. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63. Σαβισάρ Μπαχ. Πάλι με προφορική τροπολογία όπως πριν. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60 εκπίπτει. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 του κυρίου Δανέλη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 εκπίπτει 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 και 24 μαζί και υπάρχει πάλι προφορική τροπολογία την οποία βλέπετε μπροστά σας αν δεν υπάρχουν ενστάσεις τη ψηφίζουμε μαζί ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται Ακολουθεί η 25 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 με προφορική τροπολογία της εισηγήτριας χωρίς δεν υπάρχουν στάσεις υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Παραρτήματα. Τώρα τροπολογία 70 και 71 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 72 εκπίπτει. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 73 εκπίπτει. Διαιτολογικές σκέψεις 31 μπαλσάετης υπέρ κατά αποχές θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση τροπολογία 31 αρχίζει η ψηφοφορία το Λαϊκό Κόμμα έχει μία ψήφο παραπάνω κύριε Γκρός Ψηφίσατε όλοι. όχι. Βάλτε το πάλι μέσα. Έβγαλε άλλο συναδελφό σα. Πέρας. θα το επαναλάβουμε, θα την επαναλάβουμε την ψηφοφορία αυτή. Ξαναρχίζει. 31, αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι και όλες. Πέρας. «22 υπέρ 19 κατά εγκρίνεται». Τροπολογία 32. Ρίκε υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα κάνουμε και εδώ ηλεκτρονική επαλήθευση. 32 λοιπόν. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 16 υπέρ 25 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33. Για το πρώτο τμήμα, εδώ έχουμε, έχει ζητηθεί λοιπόν ψηφοφορία κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα μέχρι εκεί που λέει τροχαία ατυχήματα. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές αυτό απορρίπτεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 εκπίπτει 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ψηφίζουμε τώρα την 38 αλλά μόνο το πρώτο της μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα επαληθεύσουμε την ψηφοφορία της 36. Το κύριο Ρικέ λοιπόν. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. 28 υπέρ, 13 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 τη συγκίτρια υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 με την προφορική τροπολογία που βλέπετε μπροστά σας υπάρχουν ενστάσεις όχι καλώς ψηφίζεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία αρχίζει η ψηφοφορία με ηλεκτρονική μέθοδο ψηφίσατε πάλι μία ψήφος υπερβα... υπερβάλλουσα για το Λαϊκό Κόμμα παρακαλώ βγάλτε μία ναι, εντάξει, κάποιο έβγαλε. Τώρα βγάλατε δύο. Καλά λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 38 υπέρ, μία κατά και δύο αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Αγιάλα Σέντερ και καλή τύχη. Ας αλλάξουμε τώρα την ομάδα εδώ. Στο Προεδρείο πρόκειται τώρα για τη δική μου έκθεση για τις στατιστικές, και τις συλλογές δηλαδή στατιστικών δεδομένων. Τροπολογία 15, Μπαλσάιτης, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 19 με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία πρώτα η πρόταση όπως τροποποιήθηκε η ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει ψηφίσατε πέρας 42 ψήφοι υπέρ, χωρίς αποχές, χωρίς ψήφους κατά. Δεν τελειώσαμε ακόμη και το νομοθετικού περιεχομένου ψήφισμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας. 41 ψήφοι υπέρ, 0 και 0 κατά και αποχές. Υποθέτω λοιπόν τώρα ότι μου δίνεται την εντολή να προχωρήσω σε διαπραγματεύσεις με Συμβούλιο και Επιτροπή στην βάση του κειμένου αυτό. Καλά, γνωρίζω τις ενστάσεις της κυρίας Φώστερ. Σας ευχαριστώ λοιπόν και αν έχετε λίγη υπομονή θα πιω λίγο νερό πριν να συνεχίσουμε. Είναι και η έκθεση για τα υγρά. draft report on aviation security. Έκθεση του κυρίου Ντεγκράντε Πασκουάλ για τους σαρωτές ασφαλείας στα αεροδρόμια. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 με την προφορική αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μαζί με την προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 βαντάλεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32. Με την προφορική ενσωματωμένη, εάν δεν αντιτίθεται κανένα στις προφορικές, θα θεωρήσω ότι έχουν αναγνωστεί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά αποχές θα την ελέγξουμε την 33 Λίχτεμπεργκερ αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 20 υπέρ, 21 κατά, μία αποχή απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35. Μετά την 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 36 Λίχτεμπέργκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 wheels υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 έχει αποσύρθει πάμε στον τομέα των σαρα... σαρωτών 60 της κυρίας Λίχτεμπέργκερ 60, 84, 87, 140, 159, 167, 57 και 27 on block της ΛΥΜΠΕ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε αυτή την ομάδα τροπολογιών. Αρχίζει η ψηφοφορία. Επί αυτών των τροπολογιών που ψηφίζουμε ομαδικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 14 υπέρ, 26 κατά, απορρίπτεται. Συμβιβασμός Α. Τροπολογία συμβιβασμού Α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα 45, 43, 44, 46, 47, 48 και 49 καταπίπτουν. Συμβιβασμός Β. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται ο συμβιβασμός. Τροπολογία 50. Λίχτεμπερκερ χωριστά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε την 50. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί αλλά προτιμώ να ελέγξουμε γιατί κουραστήκατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 24 υπέρ, 18 κατά, άρα εγκρίνεται. 51 με 56 καταπίπτουν εξαιτία του συμβασμού Β, 57 για λασέντερ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 65, η 65 είναι επόμενη, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μάλλον ας ελέγξουμε την 62. Αρχίζει η ψηφοφορία, νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά καλύτερα να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 62. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 24 υπέρ, 18 κατά, εγκρίνεται. 63. Η 63 καταπίπτει, επειδή εγκρίναμε την 65. 64 τώρα. Το δεύτερο τμήμα θα πρέπει να ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Στο επόμενο τμήμα την ανάγκη αναλογικότητας 64 υπέρ, 66 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός Γ. Υπέρ. Κατά αποχές μπορούμε να ελέγξουμε τον συμβιβασμό Γ. Παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται 26 υπέρ 16 κατά. Εγκρίνεται ο Συμβιβασμός Γ. Αυτό σημαίνει 67, 68, 69, 75 μέχρι κάτω Μάλλον η 75 είναι, θα την ψηφίσουμε, είναι χωριστή. Την τελευταία πρόταση. Ποιοι είναι υπέρ της τελευταίας πρότασης, κατά αποχές απορρίπτεται. Οι άλλες καταπίπτουν 73, η τελευταία πρόταση, το points out, τονίζει υπέρ, παρακαλώ, κατά αποχές απορρίπτεται. Άρα τώρα ψηφίζουμε την 76 Λίχτεμπέργκερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά αποχές μπορούμε να ελέγξουμε παρακαλώ την 80. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 25 υπέρ, 16 κατά, καμία αποχή, άρα εγκρίνεται. 78 τσικάου υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε την 79 Γένσεν. Αρχίζει η ψηφοφορία επί της 79. Ψηφίσατε όλοι. 24 υπέρ 17 κατά. Άρα εγκρίνεται, είχατε δίκιο. 82 Wills υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 81, η 81 έχει αποσύρθει, 83 καταπίπτει, με συγχωρείτε, Αγιάλα Σέντερ, 83 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Μερικοί δεν ασχολούνται καν. Μπορούμε να ελέγξουμε την 83 Αγιάλα Σέντερ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 28 υπέρ 13 ψήφι κατά εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 88 φώστερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 με την προφορική υπέρ κατά αποχές μπορούμε να ελέγξουμε την 89 89 Μαρινέσκου αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 26 υπέρ, 15 κατά, μία αποχή, άρα εγκρίνεται. Συμβασμός Δέλτα σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, μέχρι τα δικαιώματα και αξιοπρέπεια και το δεύτερο από το τονίζει. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Από 91, 93, 92 καταπίπτουν, Φώστερ 94 υπέρ, κατά, αποχές ας ελέγξουμε. Παρακαλώ την 94 της κυρίας Φώστερ αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 29 υπέρ 12 κατά εγκρίνεται. Τρο, ε, συμβασμός ε, με συγχωρείτε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα 18, 19, 21, παράγραφοι μέχρι το, την 106, Wills, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 109. Υπέρ. Κατά απόχες απορρίπτεται. 112. Κόζα σε δύο τμήματα μέχρι η Ινσουλίνη και δεύτερο, το δεύτερο τμήμα έχει αποσυρθεί από ό,τι βλέπω. Άρα ε, ως προς την Ινσουλίνη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113. Φώστερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. J. Συμβιβασμός J. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 115, 114, 123 μέχρι κάτω καταπίπτουν μέχρι το συμβιβασμό F. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αυτές, αυτές οι ψηφοφορίες μου αρέσουν, λέει ο Πρόεδρος. 138. 139. Μπραντμπορν. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκατόν σαράντα τέσσερα. Βαντάλε μετά από την παραγραφό 3 υπέρ κα... Ας ξαναρχίσουμε. Υπέρ. Κατά αποχές μπορούμε να ελέγξουμε την 144 αρχίζει η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας 13 υπέρ 24 κατά απορρίπτεται 'Προστασία δεδομένων G' παράγραφος 27 υπέρ Το συμβασμό G κατά αποχές εγκρίνεται. 150 πενήντα Λάχτφριντ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 156 Αγιάλα Σέντερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 168 Λάιχτφριντ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην απαγόρευση υγρών. Συμβασμός L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 173, 174, μάλλον 174, Wills, υπέρ. υπέρ της 174 κατά αποχές απορρίπτεται 175 Μάισνερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 179 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε την 179 βαντάλεν αρχίζει η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας 24 υπέρ, 18 κατά, εγκρίνεται. 181 δεβεϊράκ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 182 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 184 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 183 Ψηφίζουμε την τελευταία πρόταση χρήση του ICS υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 185 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 186 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 187 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 188 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Διεθνείς σχέσεις, 189 έχει αποσυρθεί βλέπω, 109 καταπίπτει, άρα τώρα πάμε στους σαρωτές ασφαλείας, ε, τροπολογία 1 Wills υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 2 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ο συμβασμός. 14 Wills υπέρ κατά αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε την 14 σας παρακαλώ της κυρίας Wills. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 20-21 ψήφι. 15 ε, βαντάλεν υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε την 15. Υποπτεύουμε ότι θα είναι ίδιο το αποτέλεσμα και στη 15 αρχίζει όμως η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 24 υπέρ κατά 18, άρα εγκρίνεται. 16 Wills υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 Λίχτεμπεργκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19. Α, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος κάποια παρέλειψα. Με συγχωρείτε, 17 wheels υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 19 Αγιάλα Σέντερ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 καταπίπτει, 21 Λάχτφριντ, Φλέκενστάιν υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές ε, μπορούμε να ελέγξουμε την 22 της κυρίας Λίχτεμπεργκερ παρακαλώ αρχίζει η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας 20 υπέρ κατά 22 άρα απορρίπτεται 23 μπαχ υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται 24 τσικάου υπέρ κατά απόχες μπορούμε να ελέγξουμε την 24 σας παρακαλώ της κυρίας Τσικάου αρχίζει η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας 24 υπέρ 17 κατά άρα εγκρίνεται 25 wills υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στις γνωμοδοτήσεις, παράγραφος 5, γιατί πριν είχαμε συμβιβασμούς από την έμβη υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11, 12, 13, 14 μέχρι την 21 καταπίπτουν, ε, άρα την 21 πλέον ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε την παράγραφο 21, σας παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία επί της παραγράφου 21. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 20 υπέρ, 22 κατά. Απορρίπτεται. Λίμπε, παράγραφος 1, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. τρία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. τέσσερα υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί αλλά θα ήθελα να ελέγξουμε. Παράγραφος 4. Αρχίζει η ψηφοφορία επί της παραγράφου 4. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 20 υπέρ, 22 κατά. Πράγματι έχει απορρίφθει 6 ε, πολιτικές ελευθερίες υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 9. Ψηφίζουμε την παράγραφο 9 γιατί οι 7 και 8 καταπίπτουν εξαιτία των συμβιβασμών υπέρ της 9 κατά αποχές εγκρίνεται. 12, παράγραφος 12 είναι. Η επόμενη υπέρ κατά αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε παρακαλώ την παράγραφο 12. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 25 υπέρ, 17 κατά, εγκρίνεται. Παράγραφος 23 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία η οποία και αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται με 37 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 3 αποχές. Να συγχαρούμε τον κύριο Ντεγκράντες Πασκουάλ. Και τώρα συνεχίζουμε και περνάμε στο σχέδιο γνωμοδότησης για την εποπτεία της αγοράς ε, για τα δίκυκλα, τρίκυκλα και τετράκυκλα. Η συγκητής είναι ο κύριος Ζήλε. Και ξεκινάμε με την τροπολογία 4 του συγκητή. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 και 34 έχουν αποσυρθεί. Είμαστε τώρα στην τροπολογία αριθμός 5, 6, 9, 15 μαζί. Τις ψηφίζουμε. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 35 τώρα της κυρίας Τικάου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία Α. Α. Ε. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και έτσι φτάνουμε στη 14. Τροπολογία 14. Δεύτερο τμήμα. Όχι, τις 37. Της κυρίας Αγιάλα Σέντερ. Δεύτερο τμήμα της 37. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19, 20 και 21 μαζί τις ψηφίζουμε υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 7, 8, 10, 11, 12, 16 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26. Μαζί τις ψηφίζουμε όλες αυτές τις τροπολογίες. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 40-41 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τώρα. Φτάνουμε στην τροπολογία 30. Τροπολογία 30 παρακαλώ. Στο 9α. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Καταπίπτει. Καταπίπτει αν δεν έχουν εγκριθεί οι προηγούμενες, όμως εγκρίθηκαν. Πρέπει να ψηφίσουμε λοιπόν την 31. Την τροπολογία 1 πρέπει να την ψηφίσουμε. Έχετε δίκιο. Στο 3 λοιπόν, τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην 31 γιατί δύο καταπίπτει επειδή εγκρίναμε την 30. 31. Αγία Σέντερ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β. Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία τώρα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. 39 υπέρ, κανείς κατά, δύο αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Ζήλα. Καλώς. Αυτό σημαίνει ότι μετά από αυτή τη σκληρή δουλειά και την ε, μεγάλη συγκέντρωση με την οποία δουλέψαμε, τελειώσαμε για σήμερα το πρωί. Συνεχίζουμε στις 3 με την έκθεση Σερακιάνη για τον νέο Ευρωπαϊκό Συνδρομικό Χώρο. Καλό καφέ, λέει ο Πρόεδρος.